Ε, για όλη τη σημερινή συζήτηση και θα επανέλθω με τα σχόλιά τους. Βάσει του άρθρου 216 παράγραφο 4 σας ενημερώνω ότι δεν έχουν ζητηθεί να ψηφιστεί το διορθωτικό το οποίο αναγγέλθηκε σε 17 και 30. Το διορθωτικό λοιπόν θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Προχωρούμε τώρα στην ε, δήλωση της Επιτροπής